Die Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν σας έχουν διανεμηθεί. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν. Το κείμενο των πρακτικών. Ερχόμαστε στη συζήτηση επί περιπτώσεων παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία και κράτου δικαίου, καταρχά στο Αζερβαϊτζάν, ιδιαίτερη περίπτωση του Ραφίκ Τάγκη και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ ως πρώτο συντάκτη. Κύριε Πρόεδρε, η τραγική περίπτωση του Ράφικ Τάγκη είναι ένα σύμπτωμα της παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Αζερβαϊτζάν που είναι μέλος και του ΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ήταν γνωστός ε, δημοσιογράφος και δημοσίευσε ένα άρθρο που έλεγε ότι ε, η αυστηρή προσήλωση του καθεστώτος του Αλία ήταν ει βάρο της δημοκρατική πορεία της χώρας. Αποτέλεσμα, ένας ακραίος Ισλαμιστής ε, για το ΛΑΧ έβγαλε ένα φετφά και ε, τον άνθρωπο το μαχαίρωσαν και πέθανε μετά από τέσσερις μέρες. Ε, ασκήθηκε, ε, ασκήθηκε συγγνώμη, διεθνής πίεση, αλλά η κυβέρνηση της χώρας και οι αρχές δείχνουν αδιαφορία και δεν προβάλλεται πολύ η έρευνα γύρω από το θάνατό του, τη δολοφονία του. Μέχρι τώρα οι Ιρανικές αρχές ούτε έχουν καταδικάσει το ΦΕΤΦΑ, που φαίνεται ότι είναι υποκίνηση σε δολοφονία, ούτε κάνουν τίποτα για να διεξάγουν έρευνα. Ε, για να εξηχνιαστεί αυτό το έγκλημα και οι αυτοργοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Καλωσορίζουμε την απόφαση έστω και αρχή να αρισκευθεί ποινική δίωση και καλούμε τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να κάνουν ό,τι μπορούν για να οδηγηθούν οι αυτοργοί στη δικαιοσύνη ε, με δίκαιη δίκη βάσει διεθνών προτύπων. Καλούμε και τις Ιρανικές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με την έρευνα και να δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να βοηθηθεί η πορεία. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Ιράν έτσι κι δεν μας ακούει αυτά που λέμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ανησυχούμε από ότι ακούμε ότι χρησιμοποιούν το ποινικό δίκαιο στο Αζερβαϊτζάν για να εμποδίσουν τη συζήτηση για τη θρησκεία. Θα πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ελευθερία λόγου, ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις άλλες ελευθερίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Η κυρία Ντεκεζέρ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Θα ήθελα να σχολιάσω ένα κείμενο, Πρόεδρε, και να το διαβάσω. Με ναι κύρωση αυτό θα έπρεπε ο πανίσχυρος που ενέκρινε την απόφαση αυτή για να ευχαριστήσει τους μουσουλμάνους να δώσουμε να καταλάβουν μέσω αυτού του μηνύματος τους νέους ότι οι αξίες του Ισλάμ δεν ισοδυναμούν με το να επικρατήσουν οι αξίες του διεθνούς υπεριαλισμού και του σιωνισμού. Όσοι προδίδουν ε, τη θρησκεία θα πρέπει να τιμωρούνται. Και εδώ θέλω να αποτύσω φόρο τιμή στο Αζερβαϊτζάν και τον Ισλαμισμό. Αυτό δημοσιεύτηκε στο ε, ιστότοπο του Ελκαρανή μετά, την, ε, μετά το θάνατο, την ημέρα μετά το θάνατο του Ραφίκ Ταγί. Αυτό δεν είναι το Ισλάμ που θέλουμε σε αυτό το κοινοβούλιο. Και αυτή δεν είναι η πραγματική φίλη του Ισλάμ όπως αυτοί που ακούσαμε να παίρνουν το λόγο εφόσον βραβεύτηκαν το βραβείο Ζαχάροφ. Εάν ζητούμε από τις αρχές του Ιράν, του, της Μπακού, να καταδικάσουν το, την πράξη αυτή, θα πρέπει και εμείς στο Κοινοβούλιο να μην ξεχάσουμε να καταδικάζουμε με πυγμή αυτήν την, ε, αυτό το φανατισμό του Ισλάμ που μπορούμε να τον διαβάσουμε σε αυτό το κείμενο και αλλού. Θέλουμε το Ισλάμ που είναι μετριοπαθές και σέβεται της ελευθερίας σε αντίθεση με τις αρχές του Αζερβαϊτζάν και εφόσον οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν ισχύουν στην περίπτωση της δολοφονίας αυτής. Θα πρέπει λοιπόν να ε, φροντίσουμε και για την προστασία του κυρίου Σαγκάτογλου, ο οποίο ε, βρίσκεται και, και εκείνο σήμερα σε κίνδυνο για τη ζωή του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεκεζέ. Μιλήσατε ε, τόσο πολύ μέχρι να μπορέσει να πάρει το λόγο ο κύριος Σταβάρης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Ταγκή, που είναι αζέριος δημοσιογράφος και συγγραφέας, είναι ένα θύμα των συνθήκων της παγκοσμιοποίησης, ο οποίος ε, κατέκρινε δημοσίως τον ε, κύριο Αχμαντινετζάν για την προσήλωσή του στο Ισλάμ. Ο μεγάλος Αγιατολάχ, ο κύριος Γκαράνη, επικήρυξε τον Τάγκη και με τις μαχαιριές που δέχτηκε ε, δεν μπόρεσε να επιβιώσει για πολύ μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Έχει δίκιο ο Ταγκή. Το Ισλάμ είναι μια χιλιετής, ε, μια ιστορία με χιλιετή, μια θρησκεία με χιλιετή ιστορία, αλλά όχι όπως την παρουσιάζει σήμερα ο Αγιατολάχ ε, Γιακαράνη και ο, ο Πρωθυπουργό Αχμαντινέτζαν. Ουσιαστικά στιγματίζεται αυτή τη στιγμή η θρησκεία θα μπορούσε να υπάρχει συνύπαρξη του περσικού πολιτισμού με την ε, αζερική φυλή και να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη. Η Πορτογαλία λοιπόν καταδικάζει τέτοιες συμπεριφορές. Δεν... Εφόσον θα είναι μέλος και του μόνιμου, μάλλον εφόσον θα κατα... το μόνιμο συμβούλιο του ΟΗΕ από το 2012 στο 2014 το Ιράν θα πρέπει να καταδικαστεί για τα εγκλήματα που διαπράττει κατά των πολιτών της χάρος της ίδιας και άλλων εθνικότητων. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχεται τέτοιου είδου πράξει. Το συζητήσαμε και στην περασμένη σύνοδο. Υπάρχουν εταιρείε από την Ευρώπη που βοηθούν το Ιράν στην λογοκρισία του ίντερνετ, του διαδικτύου ή στον παραδημοσμό τη ελεύθερη έκφραση στο Ιράν. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να αναλάβουμε τι ευρωπαϊκέ μα αρμοδιότητε και στα ανθρώπινα δικαιώματα και αλλιώ τα λόγια μα θα παραμείνουν και ένα νοήματο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβάρες. Η κυρία Μακοβέη για ένα λεπτό παρακαλώ. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ραφίρ Τάγκη ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας στο Αζερμπαϊτζάν και είχε ασκήσει κριτική κατά της ιερανικής κυβέρνησης και της ε, θρησκευτικής καταπίεσης. Από το 2007 και μετά δεχόταν απειλές για τη ζωή του, οπότε και εκδόθηκε ο, Φετβά, ο Φετφάς. Και εκεί ζητεί το μάλιστα θάνατοσή του. Στις 23 Νοεμβρίου δολοφονήθηκε. Υπάρχουν υποψίε ότι ευθύνονται οι τοπικοί εξτρεμιστέ και η κυβέρνηση τη χώρα. Οι αρχέ εξετάζουν, ερευνούν την κατάσταση, αλλά θα πρέπει αυτή η έρευνα να είναι γρήγορη και αμερόληπτη. Και όχι μόνο οι δολοφόνοι, αλλά και όσοι διέταξαν ε, το θάνατο του, την δολοφονία του Τάγκη θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να συνεργαστεί η κυβέρνηση, να δίνοντα στοιχεία και ε, επίσης θα πρέπει οι αρχές ε, να απαγορεύσουν να ζητούν οι κληρικοί ε, ρητός ε, την ε, δολοφονία ανθρώπων. Πολλά θα εξαρτηθούν από τι θα κάνει το Ιράν πάντως. Εγώ ζητώ από τις αρχές του Αζερβαϊτζάν να κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών του Αζερβαϊτζάν και ιδίω αυτούς για τους οποίους έχει εκδοθεί φετφά. Ευχαριστώ κύριε Μακοβέη. Η κυρία Σάκε για μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Ραφίκ Τάγκη δολοφονήθηκε γιατί άσκησε το δημόσιο δικαίωμα τη ελευθερία έκφραση. Πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση και είναι πολύ σημαντικό και οι αρχέ ε, του Αζερβαϊτζάν αυτό να το πράξουν ε, με αξιόπιστο τρόπο. Επίση πρέπει το φετφά που είχε ε, εκδοθεί μετά το άρθρο που δημοσίευσε ο ο Τάγκη, ε, να δούμε αυτός ο κληρικός που τον εξέδωσε γιατί δεν τιμωρήθηκε ποτέ, γιατί δεν έχει αρθεί ακόμη. Δεν μπορεί να δίνεται άδεια για να σκοτώσουν ε, κάποιοι με, τέτοιες, ε, με Έπρεπε να είχε καταδικαστεί πολύ πιο απερίφραστα και ε, έπρεπε να, γνωρίζουμε ότι, να γνωρίζουν οι αρχές ότι κινδύνευε η ζωή του. Θα πρέπει οι αρχές του να αποφασίσουν τι είδους κοινωνία θέλουν, τι κοινωνία θέλουν να δημιουργήσουν. Η δολοφονία που μπορεί να θεωρηθεί και ένα μεμονωμένο επεισόδιο έχει λάβει πάντως χώρα ε, υποκαθεστώς μεγάλης πίεσης ότι αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα πιέζει η αντιπολίτευση και αν οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν δεν επιλέξουν να, να εφαρμόζουν όχι μόνο ε, στα χαρτιά αλλά και ουσιαστικά και τα ψηφίσματα και τις συμβάσεις ε, διεθνή και όλες τις μέσες που έχουν αναλάβει θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αντλήσει τα συμπεράσματά της. Θα πρέπει να πιέσουμε τις αρχές ε, να ακολουθήσουν το μονοπάτι προ μια πιο ελεύθερη και δίκαιη κοινωνία. Δεν είμαι βέβαια και τόσο αισιόδοξη ό,τι αφορά τη συνεργασία των Ιρανικών αρχών στο ρόλο αυτού του Ιρανού κληρικού. Όμω, ε, τουλάχιστον από τι αρχέ του Αζερμπαϊτζάν πρέπει να περιμένουμε περισσότερα και να εκμεταλλευτούμε και τι σχέσει που έχουμε με τη χώρα αυτή για να του ασκήσουμε πιέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Σάκε. Οι συντάκτε ήταν αυτοί. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Πρώτα, ε, ε, δόξα Τούνουντ Κόενστάιν. Ευχαριστώ. Ο Ραφίκ Τάγκη ήταν υπόδειγμα ελευθέρου δημοσιογράφου. Καταγόταν από το Αζερβαϊτζάν. Η οικογένειά του και μη κυβερνητικέ οργανώσεις ζητούν ε, να γίνει σωστή διερεύνηση του θανάτου του. Το Αζερβαϊτζάν είναι και μέλος της Δυτικής ε, συμμαχίας ε, και θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, γίνει σωστή η οργάνωση. Δεν μπορεί να φυλακίζονται κάποιοι ακτιβιστές που διοργανώνουν εκδηλώσεις μέσω του Facebook. Και εγώ ίδια διοργάνωσα στην Πολωνία αντίστοιχη εκδήλωση για να θυμίσω στους πάντες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε τέτοιες ε, πράξεις να ε, τιμωρούνται με φυλάκιση. Στο επόμενο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών θέλω να ε, δοθεί βραβείο μετά θάνατον στον κύριο Τάγκη για την ελεύθερη δημοσιογραφία. Κύριο Σβίγγενεν, ευχαριστώ συνάδελφοι. Αγαπη... Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω υπογράψει το κοινό ψήφισμα, αλλά θα προτιμούσα ε, το δικό μας σε έξι παραγράφους αναφέρεται το Ιράν. Δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να έχει διαφορετική διατύπωση. Είναι η τραγική περίπτωση του Ραφίκ Τάκη και δείχνει πόσο ε, μεγάλα είναι τα προβλήματα και η αλληλεξάρτηση στην περιοχή. Όταν μιλούμε για το Ζερμπαϊτζάν δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τους γειτονέ του. Έχουμε κάθε λόγο να εκφράζουμε επικρίσει για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Επανειλημμένα το έχουμε συστήσει στο Κοινοβούλιο. Αλλά θα πρέπει επίση να υποστηρίξουμε και τι αρχέ τη χώρα στην καταπολέμηση της ε, εμφάνισης ε, φονταμενταλιστών στη χώρα. Καλό την κυβέρνηση και δεν είναι εύκολο αυτό να κάνει πλήρη έρευνα και να ε, δώσει όλα τα στοιχεία στο Κοινοβούλιο. Επίσης, καλό να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για να βεβαιωθούμε ότι θα προστατευτεί ο Σαμίρ Σανταγκάτογλου, ο εκδότης που μπορεί να πέσει και αυτός θύμα των Ιρανών κληρικών. Ελπίζω αυτά τα θέματα να λυθούν πριν συνεδριάσει στον Πακού η Euronest. Ευχαριστώ κύριε Βίγκενεν. Η κυρία Βερζιά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα ευχαριστώ για τη δολοφονία του κυρίου Ταγκή. Ούτε για την κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. Αυτό το έχω κάνει ήδη στο ημικύκλιο στο παρελθόν. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω την θλίψη μου για την επιλογή στα κατεπήγοντα που έχει γίνει στην ημερήσια διάταξη και τον τρόπο που τα συζητούμε και τα εξετάζουμε. Διότι η κατάσταση των προσφύγων του Ασράφ είναι στο στρατόπεδο, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο αυτό γυναίκες και παιδιά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ανακοίνωσαν την ε, ε, την, αποχώρηση των στατευμάτων του ήδη από τον Νοέμβριο. Όμω θα πρέπει να, ληφθούν, να ληφθεί κάποια μέρημνα για τους ε, πρόσφυγες του Ασάτ. Ενώ ήδη ακόμη η κυβέρνηση του Ιράκ του θεωρεί τρομοκράτε. Κυρία Άστον, είπατε εκπρόσωπο ζήτησε προστασία για τα άτομα αυτά. Αλλά η ανώτατη, είπατε πραγματικά του ΟΗΕ, απάντησε ότι χρειάζεται χρόνο. Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη το αίτημα τη ε, κυρία Άστον, οι οποίοι έχουν και δεσμού με κάποια από τα κάτι μέλη. Θα πρέπει λοιπόν, Πρόεδρε, να ε, δούμε εδώ ότι δυστυχώ η γαλλική κυβέρνηση βρέθηκε στην πρώτη γραμμή τη υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Βεργιά. Αυτοί ήταν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ε, ο κύριος Ρέπο ζήτησε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Ραφίκ ε, Τάγκη ήταν θύμα ε, ενός φετφά από Ιρανό κληρικό λόγω των πεπιθήσεών του και αυτών που είπε. Υπήρχαν προβλήματα και τα είχε επισημάνει. πολλοί συγγραφείς, bloggers, δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ε, είναι χαλκευμένες οι κατηγορίες εναντίον τους, αλλά τους ε, κατηγορούν και τους διώκουν. Το 2013 θα γίνει μέλος ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Αζερπέτζαν, μα μπορεί μια τέτοια χώρα να εκπροσωπεί τη διεθνή κοινότητα στο σεβαστό αυτό σώμα. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να εισακωστεί. Πρέπει να υπάρξει διάλογο ε, με ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε οποιοδήποτε κράτο σέβεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσει η μισθοφόροι δολοφόνοι οι οποίοι σκότωσαν τον Τάγκη να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να ελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Ευχαριστώ. Αυτοί είχαν ζητήσει το λόγο. Ερχόμαστε στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΗ. Η κυρία Κόρχολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα ανησυχεί πολύ η κατάσταση τη δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν. Η δολοφονία αυτού του δημοσιογράφου είναι πολύ ανησυχητικό γεγονό. Και εκατοντάδε άτομα έχουν εκφράσει επικριτικά σχόλια και έχουν αντιπαραθέσει τον Ισλαμισμό με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αλλά εδώ έχουμε μια δολοφονία ως ε, συμπέρασμα. Μιλάμε για την ημέρα της διεθνούς ατιμορρησίας. Εδώ μιλάμε για δολοφονίες οι οποίες ποτέ δεν ερευνήθηκαν. Ο κυρίος Ταγκή δεν ε, έχει... Δεν πρόκειται να ερευνηθεί η υπόθεσή του, δεν πρόκειται να βρεθούν οι υπεύθυνοι. Εδώ λοιπόν χρειάζεται συστηματική δράση. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμό του όταν μπορεί κανεί να δρά κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε σε κάθε περίπτωση του υπέτειου. Ευχαριστώ κυρία Κόχολα. Η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τη λύπη μου για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Ραφίκ Τάτσι. Το καταδικάζω περίφραστα. Δείχνει που μπορεί να οδηγήσει ο θρησκευτικός εξτρεμισμός. Ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε δικαίωμα στη ζωή. Μεγάλα ερωτηματικά ανοίγει η δολοφονία αυτού του δημοσιογράφου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ζερμπαϊτζάν. Πολλό δε μάλλον μας ανησυχεί που είναι μέλος ε, και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της γειτονίας και συμμετέχει ε, ενεργά. Παρόλες αυτές τις διεθνείς σχέσεις, το Αζερβαϊτζάν δεν έχει καταφέρει ακόμα να ε, ανταποκρίνεται σοβαρά στις υποχρεώσεις του για την ελευθεροτυπία και την προστασία εκείνων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω η κυβέρνηση της χώρας να κάνει κάτι για να διερευνήσει και να τιμωρήσει ε, τους ε, αυτούργους. Θα πρέπει να σταματήσει η τιμωρησία, Διότι αυτοί οι δολοφόνοι δολοφονούν με βάση θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Θα ήθελα παρακαλώ η Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνει διαβήματα ε, στο Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κρέτσου. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω με αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Βίγκενιν. Νομίζω ότι θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να επιλέγουμε τα θέματα για αυτές τις συζητήσεις. Φυσικά και είναι λυπηρό και όλοι καταδικάζουμε αυτό που έγινε στα Αζερμπαϊτζάν. Είναι προφανές όμως ότι αυτού του είδους η κλιματικότητα δεν έχει σύνορα. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούμε για να προσπαθήσουμε στο μέλλον να αποτρέπουμε τέτοιου είδους ενέργειες που είναι ομές και βίες εξαιρετικά. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταδικάσουμε το Αζερβαϊτζάν για αυτό το δολοφονία, αλλά να ζητήσουμε από το Αζερβαϊτζάν να κινητοποιηθεί και να επιταχύνει τις ε, έρευνες για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διότι είναι σημαντικό να βρεθεί ο δράστης και αυτό είναι και αποτρεπτικό τρόπος για να αποφύγουμε στο μέλλον να έχουμε τέτοια αποτρόπια εγκλήματα. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη. Ο κύριος Πάσκα, τελευταίος από το ΚΑΤΣΙΑΙ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Αζερβαϊτζάν είναι μια χώρα φίλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθεί να εκδημοκρατήσει την κατάσταση. Ωστόσο, η Ισλαμική επιρροή των γειτόνων και κυρίως το Ιράν είναι ουσιαστική. Αυτό φαίνεται και από τη τηλεφωνία του Ραφίκ Τάτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο ενεργή σε την προσπάθειά της να πείσει και το λαό του Αζερβαϊτζάν ε, για τις δικές της αξίες, τις δικές μας αξίες. Θα πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε αυτή τη δολοφονία και να το θέσουμε υπόψη της κυβέρνησης του Ζερμπαϊτζάν για να πιστεί να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Διαδικασία κάτσε αεροκλώνεται εδώ. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Αλμούνια για να κλείσει τη συζήτηση αυτή. Εξακολουθεί να μα ανησυχεί η κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν σε τη φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε μια αυξητική τάση της καταστολής. Τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει ε, μάρτυρες πολύ σοβαρών ε, ενεργειών ε, και δράσεων των αρχών απέναντι σε διαδηλώσεις, πορείες ή απόπειρα διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων σαν αυτή τη Αραβική Άνοιξη. Ακτιβιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαδηλωτέ ε, πέφτουν θύμα επιθέσεων. Αυτό είναι λυπηρό. Και η καταστολή αυτή στην κοινότητα των πολιτών ε, συμβαδίζει με την επιδείνωση των συνθήκων για την ελευθερία έκφραση στη χώρα. Η διδέ ανεξάρτητη δημοσιογραφία φαίνεται ε, να μειώνεται, να συρρυκνούται. Έχουν παρενοχληθεί πολλοί δημοσιογράφοι κατά το παρελθόν, έχουν καταδικαστεί ε, χωρίς κατηγορίες ουσιαστικά ή έχουν δεχθεί επίθεση. Και σίγουρα ε, μέσα σε όλο αυτό το κακό πλαίσιο στις 23 Νοεμβρίου έχουμε και τη δολοφονία του Ράφικ Τάγκη. Στην πρόσφατη σύνοδο της Υποεπιτροπής ε, Δικαιοσύνης Ελευθερίας Ασφάλειας Τροπίων Δικαιωμάτων ε, του συγκεκριμένου αυτού συμβουλίου αλλά και ε, του Συμβουλίου συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν. Σε αυτέ τι ε, ευκαιρίε που μα δόθηκαν μιλήσαμε ανοιχτά στι αρχέ του Αζερμπαϊτζάν ζητώντα του να διεξαγάγουν μια μερόληπτη έρευνα και να προσαχθούν οι υπέτειοι στη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη. Πρέπει να δίνει σαφή μηνύματα για το πόσο σοβαρή είναι η υπόθεση είναι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμό για το κράτο δικαίου. Όλα αυτά είναι ακρογωνία λύθη για τη συνεργασία μας και με το Αζερβαϊτζάν. Το επίπεδο φιλοδοξίας Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχέσεων που έχει με το Αζερβαϊτζάν θα λάβει υπόψη το βαθμό στον οποίο οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται σε εθνικές πρακτικές και στην εφαρμογή των πολιτικών. Η Αντιπρόεδρος Άστον είχε τη δυνατότητα να δώσει το μήνυμα αυτό τον προηγούμενο μήνα που επισκέφθηκε τον Πακού. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω σε αυτό το πλαίσιο την κοινή δήλωση ε, του της διάσκεψης ε, της ανατολικής σχέσης που όλοι εκεί δεσμεύτηκαν να σέβονται τις αρχές της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Επίσης, ε, χαιρετίζω και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προασπίζει τις ε, θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και απέναντι στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ κύριε Αλμούνια. Έχω δεχτεί πέντε προτάσεις ε, ψηφίσματος ε, των διαφόρων πολιτικών ομάδων.